Okay, let's, let's start. Uh, λοιπόν, λοιπόν, ας... αρχίσουμε. Θέλω να σας πω πως να συνεχίσετε να μιλάτε τις γλώσσες σας. Έχουμε όλες τις γλώσσες, εκτός από τη δική μου, από το Λουξεμβούργο και γι' αυτό είμαι αναγκασμένος να μιλώ μια άλλη γλώσσα. Επειδή είμαστε λίγοι τώρα στην αίθουσα αυτή, να κάνουμε ένα σύνομο γύρο, να ακούσουμε τα ονόματά σας και από που είσαστε για να δούμε ποιος είναι εδώ. Εγώ λέγομαι το Κλωτούρμες. Είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1999 και εργάζομαι για την ιστορική αγορά, τα ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και την αποτελεσματικότητα ενέργεια. Ο συμπρόεδρο. Καλησπέρα σα. Εγώ είμαι μέλο τη Επιτροπή ε, Βιομηχανία ε, τη ε, Βουλή της Ισπανίας. Ο εισηγητής, Καλησπέρα σας είναι το παλάσιο. Γεωργιαστή από την Ισπανία, για την Ισπανία, ε, Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας. Εμείς, εμείς προεδρεύουμε, συγγνώμη, ο κύριος Λόπες είναι ο, εισηγητής, τα μπέρδεψα. Από εκεί, να αρχίσουμε από εσάς, πέστε μας ποιες είσαστε, πού εργάζεστε, είναι εκπροσωπεύετε. Ρεν Φίλιπς είναι μέλος της Ολλανδικής Βουλής εδώ, ε, Γερουσίας εδώ και τρία χρόνια. Εγώ εργάζομαι στην χημική βιομηχανία της Shell. Γιώνος Μέρας από τη Λιθουανία. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος. Καλησπέρα σας. Francesco Καζολή, είμαι γερουσιαστής στην Ιταλία, αντιπρόεδρος της ε, ομάδας ε, της PDS στην Ιερουσία, μέλος της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας. Ρομπέρτο Τόρτορη, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βιταλικής Βουλής. Ανδρέα Φρουτέρο, της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας. Σενατόρε Σαλβατόρε Τομασέλη, Κομισιόν. Επιτροπή Βιομηχανίας της Ιταλικής Βουλή, ε, Γερουσίας. Παρακαλώ. Μισά Τόμσον μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συζητική Ομάδα, Επιτροπή Βιομηχανία. Είμαι από τη Δανία εγώ. Από από την ε, Σουηδική Βουλή στο Πράσινο, Πράσινο Κόμμα. Είμαι στην Επιτροπή Βιομηχανής και Περιβάλλοντος. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, βιομηχανίας της ε, Βουλής ε, της χώρας μου. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης στη Γαλλία. Bernadette Bourset, secrétaire de la στην Γαλλική Βουλή είτε ω ε, Ευρωβουλευτή, χωρίς μικρόφωνο δυστυχώ. jméno je Alena jsem místo předsedkyně Είμαι Γαλατοσκοράδα, είμαι της στη Τσεχία. Είμαι υπεύθυνη για ευρωπαϊκά θέματα. Ράιν Βίτμαν, μέλος ε, της Βουλής Αυστρίας, ε, μέλος διαφόρων επιτροπών περιβάλλοντος, επιστήμης, άμυνας, οικονομικών και είμαι πρόσωπος επίσης ε, του κόμματός μου για την επιστήμη, έρευνα και ενέργεια. Χριστιανό Προύμα, επίσης, επίσης από το Κοινοβούλιο της Αυστρίας, πράσινη εκπρόσωπος για περιβάλλον και ενέργεια. Αυτοί είναι όλοι οι βουλευτές που είναι εδώ παρόντες, γιατί βλέπω και κάποιους άλλους στο κέντρο. Παρακαλώ. Εκπροσωπώ το Κοινοβούλιο της ε, Ρουμανίας. Είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Andis Kāpos pārstāv Latvijas Republikas Saimu. Ευχαριστώ και εγώ είμαι από τη Βουλή της Λετωνίας. Άννα Ζαλεύσκα, Πόσεου, Πόλσκα, Κομισία των Σπραφ Άννα Ζαλεύσκα από την Πολωνία, μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά είμαι και ειδική στο περιβάλλον. Πόλσκα, ε, Πόσεου, ε, ε, Από την Πολωνία και εγώ μέλος ε, του Κοινοβουλίου και είμαι και μέλος ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην ε, Πολωνική Βουλή. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. Να με συγχωρείτε. Парламента на България. Казвам се Никола Белишки σε ένα από την Βουλή τη Βουλγαρία τη Επιτροπή Περιβάλλοντο και Βιομηχανία. Μέλο τη Ελληνική Βουλή για την ενέργεια και για την Επιτροπή ε, Γεωργίας επίσης και όσον αφορά την κατανάλωση και το τρόφιμα. Κυρκινάς, μέλος της Βουλής της ε, Λιθουανίας και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Λοιπόν, ο Πρόεδρος, κατά βάση έχουμε μία ώρα. Παρακαλώ, ακούγεται η ελληνική καμπίνα. Ακούτε τα ελληνικά παρακαλώ. Εάν μας ακούτε μπορείτε να κάνετε ένα ρεύμα στην καμπίνα 7. Είμαστε στα δεξιά του Προεδρείου. Στα αριστερά. Στα... And what could potentially a community, an energy community for Europe contribute to be even more efficient on energy efficiency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 ist unbedingt nötig mit einer klaren Priorität erneuerbare Energie, damit wir auf Risikotechnologien wie Atomkraft und CCS verzichten können. Danke. Muchas gracias, Mrs. Brunner. Tenemos solicitada una palabra más y luego Mrs. Thompson ha solicitado a continuación. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Si no es así, primero Mr. Tomaselli. Después.